So, liebe Kolleginnen und Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ε, καλωσορίζω στην ε, συνεδρίασή μας. Προβλέπετε λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία σχετικά με τις ε, έρευνες ε, που διεξάγει η Όλαφ ε, σχετικά με τη συνεργασία για το γραφείο του εισαγγελέα και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Όλαφ. Συγητής είναι ο κύριος Μαρινέσκου. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Μαρινέσκου. <laughs> Er όχι, όχι, δεν έχει να πει τίποτα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η ψηφοφορία για τον τριμερή διάλογο. Θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Όποιο είναι υπέρ θα πατήσει το κουμπί, αλλά και όποιο είναι κατά επίση θα πατήσει κουμπί, αλλά άλλο κουμπί. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ich wollte auch noch ganz in Ruhe, nein, Moment, noch in Ruhe, bis die Kollegin Kretou. du musst deine Karte umdrehen. Ganz in Ruhe, lass dir Zeit. Diese halbe Minute haben wir. Alle abgestimmt? Gut, dann darf ich. Λοιπόν, ε, έκλεισε ψηφοφορία. 19 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Σας συγχαίρω ε, και σας ε, εύχομαι καλή επιτυχία στις διαπραγματεύσεις αγαπητές συνάδελφε κυρία Μαρινέσκου. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 7 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την ψηφοφορία σχετικά με την εφαρμογή των ε, διαπραγματευτικών, ε, ε, διοργανικών διαπραγματεύσεων. Εισηγητής ήταν ο κύριος Ντότς. Ψηφίζουμε επίσης με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ich schließe die Abstimmung. 19 Stimmen. 19 υπέρ, 3 αποχές, 2 όχι, άρα με μεγάλη πλειοψηφία και εδώ ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ε, διαπραγματεύσεις. Έτσι λοιπόν έκλεισε η ψηφοφορία ή οι ψηφοφορίες και πάμε στο σημείο υπερθμών 8 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την ειδική έκθεση Πρόκειται για τις ε, δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης αρκετά τα φιλόδοξης, αλλά απαιτείται η βελτίωση διαχείρισης. είναι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, η ε, είναι ο κύριος Ρινιέα που είχε ενδιαφερθεί πάρα πολύ για το θέμα αυτό από το Ρινιού. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Νικόλαο Μιλιώνη. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Uh, Madam Chair, honorable members of the European Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που μα προσκαλέσατε στη σημερινή συνεδρίαση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να είμαι εδώ σήμερα για να παρουσιάσω την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου για την διασυνοριακή πρόσβαση στην υγειονομική περιθέλεψη. Μέχρι πρόσφατα, ο κύριος Βασιτσόφσκι ήταν το μέλος που υπέβαλε εκθέσεις, εγώ τον αντικαθιστώ σήμερα εδώ. Ενώ η υγειονομική περίθαλψη εν γέννη χορηγείται στο εσωτερικό κάθε χώρα σε κάποιε περιπτώσει η πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για την υγειονομική περίθαλψη ενό ασθενού βρίσκεται σε άλλο κρατό μέλο. Η βελτίωση λοιπόν τη ε, διασωνηριακή πρόσβαση και αποτελεσματικότητα τη υγειονομικής περίθαλψη είναι ένα τομέα στον οποίο η ευρωπαϊκή δράση μπορεί να επιφέρει προστατευμένη αξία για του πολίτε. Η οδηγία του 2011 για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έχει ως στόχο να διασφαλίσει το δικαίωμα των Ευρωπαίων ασθενών στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ε, πέρα από σύνορα και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σε ένα φάσμα τομέων. Μεταξύ άλλων, η ανταλλαγή διασυνοριακά των ε, δεδομένων των ασθενών και η πρόσβαση ε, των ασθενών σε γενομική περίθαλψη σε περιπτώσεις ε, σπανίων ασθενών και νόσων. Δυστυχώ όμω υπάρχουν ε, προκλήσει σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε άλλε χώρε. Μόνο μικρό αριθμό μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζουν τα δικαιώματά του σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή νομική περίθαλψη. Ε, ο έλεγχο μα επικεντρώθηκε στην οδηγία λοιπόν αυτή. Δεν καλύψαμε τον κανονισμό για τον συντονισμό των ε, συστημάτων κοινωνική ασφάλισης που σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με τις ε, αναπάντεχες θεραπείες, δηλαδή τι μη προγραμματισμένες θεραπείες, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Η χρήση λοιπόν και η υλοποίηση της, εφαρμο... της οδηγίας ποικίλει μεταξύ των κρατών μελών. Στη Γαλλία είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό των ασθενών 150.000 ασθενείς περίπου το 2016 και στη συνέχεια είχαμε Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο ε, που σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ασθενών που δέχονταν στην επικράτειά τους. Στον έλεγχο λοιπόν αυτών ελέγξαμε κατά πόσο οι ευρωπαϊκές ενέργειες ε, έχουν τα απαραίτητα ωφέλη για τους ασθενείς. Διενεργήσαμε τον έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, διενεργήσαμε ε, επισκέψεις ε, συλλογής στοιχείων σε πέντε κρατημέλη, Δανία, Ιταλία, Λιθουανία, κατοχώρες και Σουηδία. Το συμπέρασμά μας συνολικά είναι ότι ενώ οι ευρωπαϊκές ενέργειες στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ήταν φιλόδοξες και βελτίωναν ε, τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, απαιτούσαν καλύτερη διαχείριση. Ο αντίκτυπος του ασθενείς ήταν περιορισμένος κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά παρακολούθησε την υλοποίηση τη ε, οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Στήριξε το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφή που ήταν αρμόδια για την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά του. Ωστόσο, κάποιες φορές ε, είναι δύσκολο για τους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη ενημέρωση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ε, σπάνιες νόσους. Η πολυπλοκότητα του πλαισίου καθιστά δύσκολη και την καθαρή ενημέρωση και ορθή ενημέρωση των ασθενών. Κατά τη στιγμή διενέργειας του ελέγχου, τον Νοέμβριο του 2018 δηλαδή, τα κράτη-μέλη μόλις άρχισαν να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ασθενών, όπως οι συνταγές, συνταγογραφήσεις, ε, ιστορικά των ασθενών κτλ και έτσι τα ωφέλη ε, αυτής της διασυνεργική δεν μπορούσαν να καταδειχθούν. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε καλύτερα να έχει προγραμματίσει την υλοποίηση της νέας της στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία, e-health strategy, ε, και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες ε, σε ό,τι αφορά ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα ηλεκτρονικής υγείας. Επιπλέον, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πιθανή ε, υλοποίηση αυτών των ανταλλαγών για ήταν υπερβολικά αισιόδοξε. Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές ενέργειες για τις σπάνιες νόσους, ε, τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς είναι μια φιλόδοξη καινοτομία και την χάνουν ευρεία στήριξη από τα διαφορετικά μέρη μεταξύ 27 και 36 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από σπάνιες νόσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ε, καταγράψει την πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει στην υλοποίηση της στρατηγικής για τις σπάνιες νόσους από το 2014. Η διαδικασία θέσπισης ε, των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς ε, στιγματίστηκε από ελλείψεις και αδυναμίες. Τελικά, υπήρχε μια πρόκληση σε ό,τι αφορά την διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και της δυνατότητας ε, λειτουργίας εντός και ε, μεταξύ εθνικών ε, συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Με βάση αυτά τα συμπεράσματα, συστήνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει καλύτερη κατεύθυνση και καθοδήγηση προς τα εθνικά σημεία επαφής για την βελτίωση της ενημέρωσης προς τους ασθενείς, να βελτιώσει και να προετοιμάσει καλύτερα τις διασυνοριακές ανταλλαγέ ε, δεδομένων υγείας, να βελτιώσει τη στήριξη και την διαχείριση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς για να διασφαλίσει, να διευκολύνει την πρόσβαση ε, σε ασθενείς με σπάνιες νόσους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και βεβαίω με τα χαράς να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ο λόγος στον Κριστιαν Γκίνια, σκιώδη εισηγητή. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στον κύριο Μιλιώνη και στην ομάδα του για την πολύ καλή δουλειά. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα μόλις εκείνος ανέφερε. Ουσιαστικά η οδηγία του 2011 ήταν ε, σημαντικό βήμα για τους Ευρωπαίους ε, ασθενείς που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε διασυνοριακή περίθαλψη. Χαιρετίζω την έκθεση, τα εν γέννη θετικά συμπεράσματα. Θα ήθελα επίση να πω ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των προσδοκιών που δημιουργήσε η υιοθέτηση αυτή τη οδηγία και του τελικού αντικτύπου, τον, του πραγματικού αποτελέσματο για του ασθενεί. Και αυτό είναι ένα παράδοξο. Έχουμε καλά συμπεράσματα, όμως η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Και τώρα ερμηνεύω λίγο εδώ την έκθεση. Τα κράτη-μέλη φέρουν το μεγαλύτερο κομμάτι της ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Πρέπει να αυξήσουν ε, τις ε, προσπάθειές τους για τα δικαιώματα των ασθενών. Μια μικρή μειονότητα μόνο των ασθενών, ε, των Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, κάτω του 20%. Και πάλι υπάρχουν δυσκολίες ότι αφορά την ανταλλαγή διασυνοριακά των ε, στοιχείων μεταξύ κρατών μελών. Πρέπει να αυξηθούν και να τεθούν οι προσπάθειες για ε, τις ε, ψηφιακές υποδομές για την υγεία. Είναι κάτι το οποίο έχουμε θίξει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Χαιρετίζω την έκθεση και θα στείλω και τις παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Vielen herzlichen Dank. Es hat sich zu Wort gemeldet. Η Κατερίνα Κινίτσι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δόκτωρα Μιλιώνη για την παρουσίασή του ε, που μας έδωσε και κάποιες ε, πληροφορίες ε, πολύ πλήρηση και κατά κάποιο τρόπο απήντησε και σε ερωτήσεις που είχα σκοπό να κάνω ε, και που με οδηγεί και στην παρατήρηση που έκανε ο προλαλής σας συνάδελφος, δηλαδή ότι το σύστημα είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον, που όμως δυστυχώς δεν παράγει τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσαμε, υποστηρίζοντας ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και που ζητούν πρόσβαση σε διασνοριακή περίθαλψη. Ε, εγώ λοιπόν ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι έκανε η Κομισιόν ε, πέρα από τις πληροφορίες που ήδη βλέπουμε και τι μπορεί να κάνει έτσι ώστε να ε, αυξηθεί η γνώση των πολιτών, η ορατότητα δηλαδή αυτού του συστήματος, να ξέρουν οι πολίτες ότι μπορούν να προστρέξουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας διασυνοριακά. Επίσης, να ρωτήσω, υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία πιο εξειδικευμένα τα οποία να υπογραμμίζουν ακριβώς ε, την διαφορά όσον αφορά την επίπτωση στην ε, υγεία, δηλαδή πια ε, κάποιες επιπλέον πληροφορίες για αυτούς που καταφέρνουν να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα περίθαλψης και αυτούς που δεν τα καταφέρνουν. Αναφέρομαι κυρίως εδώ στις σπάνιες ασθένειες. Επίσης, μια μικρή αναφορά στην χρηματοδότηση σε αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης ε, του δικτύου REN ή Κομισιόν σε σχέση με όσα ακούσαμε θέλει ή Κομισιόν σε σχέση με, και σύμφωνα με όσα ακούσαμε, ε, θέλει η Κομισιόν, λέω, να απλοποιήσει αυτήν την χρηματοδοτική υποστήριξη ποιοι θα είναι οι όροι αυτή τη απλούστευσης, θα είναι χρήσιμη αυτή η απλούστευση. Και μία τελευταία ερώτηση πριν σταματήσω σε σχέση με τα συστήματα τα οποία έχει αναπτύξει η Κομισιόν επί τη βάση της οδηγίας κυρίως ΔΕ ή κυρίως βάσει του δικτύου ΡΕΝ ε, και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τις ε, ε, κλινικές καρτέλες. Ε, λόγω της περιπλοκότητας του συστήματος ε, τίθεται και ζήτημα ε, privacy, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ρωτώ λοιπόν αν είσαστε σε θέση να μας πείτε κάποια στοιχεία παραπάνω σχετικά με τα όσα έκανε η Κομισιόν και σχετικά με το κατά πόσον η Κομισιόν μπορεί να ελέγξει το σεβασμό της προστασίας των, προσωπικών ε, δεδομένων. Ξέρουμε ότι υπάρχει και το κυβερνοέγκλημα, ξέρουμε πόσο εύκολα μπορεί να προκύψει τέτοιου είδους ε, εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, εκεί δηλαδή που ανταλλάσσονται τα στοιχεία. Γι' αυτό θα θέλαμε να μας δώσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες και οπωσδήποτε σας ευχαριστούμε και για την παρουσία σας εδώ, αλλά και για την εργασία την οποία έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, δεν βλέπω να επιθυμεί κανείς το λόγο. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, που εκπροσωπείται βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ο Διευθυντής κύριος Ρης ε, και παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την έκθεση και ευχαριστούμε και τον εισηγητή για όλα αυτά που μας είπε. Αλλά ε, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η ειδική έκθεση μας βοήθησε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, που πρέπει να βελτιωθούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι σε ορισμένε τομεί ε, λειτουργήσαμε προδραστικά, παραδείγματο χάρη όσον αφορά όλα τα ε, εθνικά σημεία επαφής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Κυρίως το δικαστήριο ζήτησε να διασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ε, προσπελασιμότητα με τους ε, ειδικού στα εθνικά σημεία επαφής. Όπως ε, βλέπετε και από την έκθεση, εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τα εθνικά σημεία επαφής. Βεβαίω έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά. Ακόμα πολλά μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω. Η έκθεση αναφέρει ότι ε, θα πρέπει να δημοσιευτεί ένα εγχειρίδιο, το οποίο μεταξύ ήδη δημοσιεύτηκε και εμείς ε, θα μεταφράσουμε το toolbox σε όλες τις ε, ευρωπαϊκές γλώσσες. Γιατί ο γλωσσικός φραγμός είναι ένα θέμα που και αυτό συζητήθηκε. Ε, εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα καθεστώς πολυγλωσσικό ε, και στα 24 δίκτυα. Είναι σημαντικό όταν οι ασθενείς αναζητούν κάποια θεραπεία ή κάποιες πληροφορίες να μπορούν να τις βρουν στη γλώσσα τους και αυτό ισχύει όχι μόνο για τους ασθενείς αλλά και για τους γιατρούς. Επίσης ε, έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα ελέγχου Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου που έχει καθερωθεί και παράλληλα προσφέρουμε μία συγκεκριμένη πρόταση για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είμαστε σε διάλογο με τα κρατημέλη για την ε, επαφή από τις διάφορες χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να προσφέρουμε ε, κονδύλια, αλλά ε, την ίδια στιγμή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έρθουμε και σε επαφή σε ε, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα στην ε, ενωσιακή, στην ευρωπαϊκή αναφορά, τους συντονιστές είναι άτομα που προείστανται, που συνεργάζονται ως ομάδα ένα από τα βασικά θέματα που μας αφορά τουλάχιστον για φέτος είναι η εισαγωγή εισαγωγή του ΡΕΝ στο εθνικό σύστημα. Αυτή είναι ε, η βασική μας δουλειά, το πρωτορχικό μας καθήκον για τα επόμενα χρόνια. Ε, βέβαια, η ε, υγεία και η προστασία της υγείας ε, παραμένει ένα θέμα σε εθνική αρμοδιότητα στα χέρια των κρατών μελών. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ψηφιακή θεραπεία. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο ότι έχουμε πολύ αναπτυγμένα προγράμματα, αλλά χωρίς τη βοήθεια των κρατών μελών και των ε, περιφερειακών ε, κυβερνήσεων, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε. Όσον αφορά τώρα ε, την ψηφιακή υποδομή για την ηλεκτρονική αντιμετώπιση της υγείας, αυτό είναι ένα πολύ περίπλοκο και προχωρημένο σύστημα, αφορά την ελεύθερη μετακίνηση ατόμων, επιτρέποντας στους γιατρούς ή στους φαρμακοποιούς ε, να μπορούν να επικοινωνούν στη δική τους ε, τη γλώσσα. Ε, θα μπορούσε ας πούμε, κάποιος να γράψει τα ιταλικά και αυτό να το διαβάζει κάποιος άλλος στα γαλλικά, στο Βέλγιο ή στη Γαλλία. Θα ήθελα να εξηγήσω ακριβώς ε, στην ερώτηση που θέσατε και ορισμένα άλλα θέματα. Όσον αφορά τους αριθμούς, όταν έγινε η έκθεση, το σύστημα ήταν ακόμα σε προετοιμασία. Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν να δημιουργηθεί, να επικρατήσει ένα είδος αξιοπιστίας στα κράτη-μέλη, ένα σύστημα σταθερό, να είναι ασφαλές, να προβλέπει την προστασία των δεδομένων. Ε, βεβαίως ε, το σύστημα είναι αρκετά αργό εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτημα των κρατών μελών έχουμε τη δική μας την υπηρεσία ελέγχου για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν εμπιστοσύνη ανάμεσά τους. Σήμερα όμως μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η πρώτη ανταλλαγή μεταξύ ε, Φινλανδίας και Εστονίας ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου και μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 6.000 ε, συνταγές που προέκυψαν μέσα από αυτό το σύστημα. Οι ασθενείς πηγαίνουν από την Εστονία στη Φινλανδία, μπορούν εκεί να αποκτήσουν ε, τα φάρμακά τους ε, και αυτό νομίζω ότι είναι μια μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη. Η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Πορτογαλία ε, προβλέπεται να περάσουν στη φάση παραγωγής πολύ σύντομα. Λουξεμβούργο, Τσεχία και η Κροατία άρχισαν ε, να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικές συνταγές και ιστορικό ασθενών. 22 κράτη θα αρχίσουν τις ανταλλαγές μέχρι το 2022 και ελπίζουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα προσχωρήσουν σε αυτό το σύστημα και η Νορβηγία. Ε, επίσης, θα θέλαμε να προσθέτουμε εικόνες, ε, τα αποτελέσματα εργαστηρίων, επιστολές. αυτά μέσα στο πρόγραμμα που έχουμε ε, συστήσει για να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό ιστορικό ασθενούς. Και αυτά όλα για να έχουμε ε, να μπορούμε να πείσουμε τους επαγγελματίες να συνεργαστούν και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα. Το ελεκτικό συνέδριο ε, χαιρετίζει την εφαρμογή, τον έλεγχο της οδηγίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με αυτή την τόσο σημαντική ε, οδηγία. Ε, καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες μέχρι τώρα. Και θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι δεν είναι ότι είμαι εγώ μόνος διευθυντής, αλλά έχουμε μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει πάνω σε αυτό και έχουμε να αντιμετωπίσουμε 28 διαφορετικά συστήματα. Άρα δηλαδή κάθε φορά πρέπει να μεταβούμε επιτόπου στο κράτος μέλος για να δούμε πώς μπορεί να γίνει βέλτιστη εφαρμογή της οδηγίας. Είμαστε σε συζητήσεις ε, με κάποια κράτη-μέλη, ε, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξελόγησή μας, γιατί είναι πολύ περίπλοκα τα εθνικά συστήματα και η διασύνδεσή τους με την οδηγία. Ε, κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε κατά τους επόμενους μήνες να ολοκληρώσουμε αυτήν την εργασία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω ε, σε αυτή την πρόταση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, πολλοί έλεγχοι θα βοηθήσουν την ε, Κομισιόν να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να έχουν καλύτερη προσφορά θεραπείες σε ασθενείς όταν βρίσκονται σε διαφορετικό κράτος μέλος. Θέλω να πω επίσης τα εξής όσον αφορά τη συνειδητοποίηση. όσον αφορά την ε, ε, ευαισθητοποίηση. Το 2014 έγινε μία μελέτη και συζητήσαμε το ότι πρέπει να επαναληφθεί εν ευθέτω χρόνο όλη αυτή η πρακτική γιατί πρέπει να δούμε ε, ποιο ακριβώς είναι το αποτέλεσμα των εξελίξεων, τα σημεία επαφής, εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχουμε δυνατότητες επικοινωνίας, αλλά έχουμε και τα όρια μας. Ε, είδαμε ότι τα κράτη-μέλη, οποτεδήποτε επένδυσαν στην επικοινωνία, είδαμε ότι ε, πολλοί πήγαν στα σημεία επαφής, πήγαν για να πάρουν τουλάχιστον πληροφορίες. Το επόμενο ερώτημα που ήταν πώς ακριβώς αλλάζει το θέμα της ευαισθητοποίησης. Αυτό το δίκτυο, το ευρωπαϊκό δίκτυο, από τότε που ξεκίνησε, επιτρέπει το να ε, μεταφέρει τη γνώση και να μην πρέπει να μετακινείται ο ασθενής. Είμαστε υπερήφανοι για την πλατφόρμα. Ε, είναι αρκετά καινοτόμα, Έχουμε δύσκολους ασθενείς, περίπλοκες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη στη Σόφια. Ο γιατρός στη Σόφια αποφάσισε αυτόν τον ασθενή να τον ε, παρουσιάσει σε έναν από τους ε, καλύτερους που ε, μπορεί κανείς να βρει σε αυτό το εικονικό τραπέζι στην Ευρώπη. Οι καθηγητές, οι γιατροί συζητάνε ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης του ασθενούς. Καταρχήν η διάγνωση, μετά συζητιέται η θεραπεία και μερικές φορές συζητάνε και άλλες επιλογές τα αν όχι θεραπεία, να προσφέρουμε καλύτερη περίθαλψη, αποκατάσταση. Αυτά συμβαίνουν. Έχουμε λοιπόν πάνω από 700 τέτοιες ε, περιπτώσεις που προέκυψαν τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, μπορούμε να πούμε ότι κάθε μέρα ε, τουλάχιστον ένας ασθενής περνάει μέσα από το σύστημα και μπορεί κανείς να διορτηθεί. Είναι ικανοποιητικό ο αριθμός. Παροχή συμβουλών είναι κάτι το περίπλοκο, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει κανείς ως γιατρός να αποφασίσει εάν υπάρχει τέτοια δυσκολία που να θέλει να απευθυνθεί σε άλλους γιατρούς. Το επόμενο είναι να υπάρχει καλή επιλογή των γιατρών και το τρίτο είναι ότι ό,τι προκύπτει από αυτές τις συζητήσεις να φτάσει στον ασθενή ο επόμενος ασθενής ε, μπορεί να μην χρειαστεί όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν έχουμε δεδομένα για το ε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την περίθαλψη, τη διάγνωση των ασθενών, αλλά γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι σημαντικό ε, να συνεργαστούν κλινικοί γιατροί και τώρα αρχίζουμε να θεσπίζουμε κλινικές οδηγίες. Υπάρχει συνεργασία, επικοινωνία μέσα από τα δίκτυα, μέσα από άλλες πλατφόρμες. Γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών, ψηφιακά εργαλεία εκμάθησης. Ελπίζουμε, αν λειτουργήσει όλο αυτό το κόνσεπτ, η γνώση θα πάρει καλύτερα αποτελέσματα στο μεμονωμένο ασθενή. Και όπως σας είπα, το κόνσεπτ είναι ε, να ε, μετακινείται η γνώση και όχι ο ασθενής. Υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο το να επιτρέπεται οι γιατροί να ταξιδεύουν για να αποκτήσουν τη γνώση. Έχουμε ένα νέο project που θα εμφανιστεί σύντομα στην αγορά και θα ε, ε, επιτρέπει, δίνω και πάλι ένα πρακτικό παράδειγμα, ο νευροχειρούργος από τη Λιόν να μπορεί να μεταβεί στη Ρουμανία ή στη Γερμανία και να χειρουργήσει ε, μία ή τέσσερις εβδομάδες από κοινού με άλλους συναδέλφους σε ένα νοσοκομείο και ε, παράλληλα κάποιος άλλος γιατρός να πάει στη Λιόν και να μάθει πώς αντιμετωπίζονται ε, περίπλοκες ε, περιπτώσεις. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά ε, για να μετακινείται η γνώση ε, μαζί με το γιατρό. Η απλοποίηση των πληρωμών τώρα έχει να κάνει με τους ασθενείς. Πώς δηλαδή θα αποζημιώνεται ο ασθενής από το σύστημα. Και πάλι αυτό να αναπόκειται στα κράτη-μέλη. Ένα από του στόχους μας για τις αρχές του επόμενου έτους είναι να βελτιώσουμε αυτήν την κατάσταση. Γιατί τα ξέρουμε, τα συζητάμε, δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζουμε. Ελπίζουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι πραγματικά τα εμπόδια, γιατί συχνά δεν είχαμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Γιατί τελικά βλέπουμε ότι εκατομμύρια ασθενεί μετακινούνται, αλλά όλοι προτιμούν να την χάνουν θεραπεία στη χώρα τους. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, αυτό ευρύτερα ισχύει. Είναι σημαντικό λοιπόν να έρονται τα προσκόμματα. Δεν έχω απάντηση θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά εμεί σίγουρα θα συνεχίσουμε να το συζητούμε με τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, μίλησα για την προστασία δεδομένων, για την ανταλλαγή στοιχείων. Οριστικοποιούμε τώρα την αναθεώρηση της εκτελεστικής πράξης, που είναι ως εργαλείο για τα κράτη-μέλη. Βρισκόμαστε στα τελικά βήματα υιοθέτηση από την ε, Κομισιόν που θα μας δώσει τα καλύτερα δυνατά μέσα προστασίας ε, του ιστορικού των ασθενών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Διευθύντα Ρή. Μας δώσατε μια πάρα πολύ καλή γενική εικόνα. Δεν ξέρω αν κάποιο από του συναδέλφου. θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο. Από ό,τι βλέπω όχι. Ως εκ τούτου θα ήθελα να δώσω το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον ε, κύριο Νικόλαο Μιλιώνη, ο οποίος ήρθε σήμερα για αυτή την ειδική έκθεση σήμερα στο Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, εν συνόψη ε, να πω ότι στην δική μας ε, έκθεση βλέπουμε, διαπιστώνουμε ε, πρόοδο σε κάποιους τομείς της υλοποίησης της οδηγίας. Ωστόσο, πολλή δουλειά παραμένει να γίνει από τη μεριά της Κομισιόν ε, και βεβαίως υπάρχει ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης των δυσκολιών που έχουμε αναφέρει Επίσης, ε, καλό είναι να υπάρξουν ε, επιπλέον πληροφορίες και input ε, που επικοδομητικά θα βοηθήσουν την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Άλλη μια φορά, αν θέλει ο κύριος συγητής να πάρει το λόγο. Representative of the Commission for the details. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά και ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Ε, αυτό το παράδειγμα της Φιλανδίας και της Εσθονίας ε, πραγματικά με εντυπωσίασε. Μακάρι ε, τέτοιου είδους συνεργασίες ε, να γίνονται και σε άλλες χώρες και ελπίζω ότι και η χώρα μου η Ρουμανία θα μπει σε αυτή την πλατφόρμα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Η πλατφόρμα bringt wirklich einen europäischen Mehrwert, Νομίζω ότι η πλατφόρμα αυτή προσφέρει ευρωπαϊκή υπεραξία, όπως το λένε έτσι πολύ κομψά και πολύ συμπαθητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι περνάμε στο υπαριθμό 9 σημείο τη σημερινή διάταξη. Είναι έκθεση υπαριθμών 12 του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, πρόκειται για το ηλεκτρονικό εμπόριο πολλές από τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ίσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνιακών δεσμών δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Ε, πρόκειται για μια ειδική έκθεση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλές απάτες στο ΦΠΑ, στους ε, δασμούς. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ε, μπορώ να καλωσορίσω τον Ιλντικό Καλ Πέλτ σε αυτήν την ε, επιτροπή. επόμενο θα λάβει το λόγο ο κύριο Ντόιτς ε, γιατί είναι ο εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πάντα με μεγάλη χαρά έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήρθα εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω την ειδική μας έκθεση όσον αφορά τις προκλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως όσον αφορά τον ΦΠΑ και τους ε, τελωνιακούς ε, δασμούς. Ας ξεκινήσουμε απευθείας με την πρώτη διαφάνεια. Τα, πρώτα σημεία, τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής. η μεθοδολογία, το εύρος ε, του, του ελέγχου του ε, audit και προχωράμε λοιπόν. Ε, ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα τμήμα του εμπορίου που αυξάνεται, διευρύνεται όλο και περισσότερο. Αλλά για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε έναν καλό χώρο ηλεκτρονικού εμπορίου προς όφελος όλων, θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες προσαρμογές που άλλωστε έχουν αναφερθεί ήδη σε άλλες διαδικασίες ελέγχου audit και όσον αφορά τους τελωνιακούς δασμούς και όσον αφορά τον ΦΠΑ. Ε, αυτά τα στοιχεία παρουσιάζουν μεγάλες προκλήσεις ε, όσον αφορά την, ε, το πεδίο νομικής εμβέλειας και δυνατότητα παρέμβασης θα πρέπει να δούμε εάν και κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις προκλήσεις. Το πεδίο εφαρμογής και τα κριτήρια, ε, καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα, από συγκεκριμένα κράτη-μέλη και την Κομισιόν ε, ήταν τα στοιχεία τα οποία ε, ελέγξαμε. Ε, σε σχέση ε, και με τα μικρά δέματα, μικρές αποστολές, ε, επίσης και οτιδήποτε σχετίζεται με την εννέα θηρίδα, την, τον όγκο των δηλώσεων που έχουν καταθέσει οι εμπορευόμενοι στο δικό τους κράτος μέλος και σε άλλα κράτη-μέλη μαζί με τις ε, αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την Κομισιόν δουλέψαμε έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε αυτόν τον οικονομικό έλεγχο ε, και ξεκίνησε η περίοδος ελέγχου από την αρχή του 2015 μέχρι και το τέλος του 2018. Εδώ σας δείχνω σε αυτή τη διαφάνεια κάποια από τα ευρήματά μας, τα οποία χωρίζουμε σε τέσσερις κατηγορίες. Πρώτον, προέκυψε ότι τα κράτη-μέλη δεν εκμεταλλεύονται τις ρυθμίσεις ε, πλήρως, τις ρυθμίσεις ε, της διοικητικής ε, συνεργασίας, καθώς επίσης και της αμοιβαίας διοικητικής αρρωγής. Επίσης ε, υπάρχουν ε, ζητήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Ε, αναγνωρίστηκε ότι τα κράτη-μέλη δεν βρίσκουν εύκολα τις πληροφορίες ανεβασμένες στο διαδίκτυο. Και εδώ είναι και οι συστάσεις συστήνουμε στην Κομισιόν να παρακολουθεί εκτενώς ε, εάν και κατά πόσον οι τρίτες χώρες, μη ευρωπαϊκές, ε, μη, μη ενωσιακές ε, χώρες ανταποκρίνονται στα αιτήματα τα οποία έχουν στείλει τα κράτη-μέλη. Επίσης, να χρησιμοποιήσουν δομές και πλαίσια τα οποία έχουν ληφθεί στα πλαίσια αυτών των ειδικών συμφωνιών για την ανταπόκριση σε συγκεκριμένες προκλήσεις. Επίσης, ε, βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερο συντονισμός ε, με τις διαδικασίες και κλπ. Επίσης, Ε, ένα από τα ευρήματα είναι ότι τα κράτη-μέλη μέσω των αρχών τους των φορολογικών δεν κάνουν εκτενείς ε, ελέγχους ούτε και η Κομισιόν ε, και επίσης ότι δεν γίνονται αρκετοί έλεγχοι όσον αφορά τις αποστολές μικρής αξίας για τα στοιχεία αυτά εμείς προτείνουμε να γίνονται περισσότερες επιθεωρήσεις από τα κράτη-μέλη καθώς επίσης ε, και κυρίως ε, όσον αφορά την απαλλαγή των μικρών, μικρής αξίας αποστολών καθώς επίσης ε, και να παρακολουθείτε η λειτουργία των από εξαποστάσεως πολίσεων. Δυστυχώς υπάρχουν ε, και κάποια ε, ζητήματα ε, όσον αφορά κάποια είδη πληρωμών και κυρίως όσον αφορά την συμμόρφωση με τις αρχές του ΦΠΑ και τα όσα μέχρι τώρα εφαρμόζονται δεν έχουν δώσει τα, τα απαραίτητα αποτελέσματα. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις πληρωμές ΜΟΣ. Ε, για τα ευρήματα αυτά εμείς προτείνουμε να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να δημιουργήσουν την σωστή μεθοδολογία ε, για ε, να μπορέσουν να κάνουν περιοδικές αξιολογήσεις της συμμόρφωσης όσον αφορά το έλλειμμα του ΦΠΑ και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όσον αφορά τώρα το ρυθμιστικό πλαίσιο και σύστημα, ε, εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις. Φαίνεται ότι οι νέες ε, διατάξεις έχουν αντιμετωπίσει ε, κάποιες δυσκολίες ή προβλήματα του παρόντος πλαισίου. Αυτές οι νέες δηλαδή διατάξεις οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ το 2021 ε, και είτε πρόκειται για σχέσεις από Ευρω... χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλη χώρα μέλος είτε πρόκειται σε σχέσεις με τρίτες ε, χώρες. Η Κομισιόν έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα ε, που διευκολύνει τις διαδικασίες από ε, τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης ε, και, του, και για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το σύστημα ε, συλλογής, το σύστημα πληρωμής βάσει ενός technology-based συστήματος. Επίσης, ε, το νομοθετικό, το εθνιστικό πλαίσιο ακολουθεί τις διεθνείς καλές πρακτικές έτσι όπως αυτές έχουν καταρτιστεί από τον ΠΟΕ και από τον ε, ΟΣΑ. Ε, και εδώ φτάνω και στο τελευταίο, στην τελευταία μου διαφάνεια ε, και το Κοινοβούλιο άλλωστε στην έκθεση TAX 3 προτείνει στην Κομισιόν ε, να ε, βελτιώσουν την χρήση των συστημάτων και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πληρωμών ε, και να συμπεριλάβουν και την χρήση των ψηφιακών νομισμάτων, καθώς επίσης να αντιμετωπίσουμε τον τρόπο αυτό και την απάτη ΦΠΑ ε, στο ε, ηλεκτρονικό εμπόριο. Οπωσδήποτε θα πρέπει τα κράτη-μέλη διαρκώς να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των εμπορευομένων των κρατών μελών με αυτό το όριο των 10.000 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πράγματι νομίζω ότι αυτό το εμπόριο είναι ένα από τα σημαντικότερα που εξετάζουμε εδώ στη δική μας την Επιτροπή και γι' αυτό αυτή η δική έκθεση είναι για μας πολύ σημαντική. Και ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας Ντότς, ο οποίος είναι συγητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα όχι μόνο να περιστώ στα συνήθι ευχολόγια και στις ευχαριστίες ε, προς την κυρία Ιντικο Γκαλπέλς. Είναι μία έκθεση που έχει ε, συνταχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ όμως, ε, διότι εντωμεταξύ υπήρξαν και αρκετές άλλες ε, ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, εκθέσεις ε, οι οποίες έτυξαν εξίσου σημαντικά θέματα. Θέματα επί των οποίων πραγματικά πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Είμαστε ειδικοί του ηλεκτρονικού εμπορίου, εμείς ε, έχουμε αγοράσει από το ηλεκτρονικά ε, εισιτήρια κυματογράφου, σαντιγή, πάρα πολλά. Ε, γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είμαστε ειδικοί του ηλεκτρονικού εμπορίου. Βεβαίως δεν θέλω να περιστώ σε αστεία, σε διάφορα αστεία περιστατικά. Θέλω να πω ότι η ψηφιοποίηση εξελίσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και η ψηφιοποίηση έχει πολλές ε, προεκτάσεις. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ε, στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο. Η έκθεση ήταν ιδιαίτερα ενημερωτική, Έχουμε 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι και οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αν τις δούμε όλες μαζί, καταλήγουμε στο ότι περίπου το 20% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη προσφέρουν τα προϊόντα τους ηλεκτρονικά. Ε, και βεβαίως ε, ε, ο όγκος ποικίλει. Πρέπει όμως ε, να έχουμε κατά νου ότι βασικά αυτό το θέμα δεν, είναι, δεν εμπίπτει απόλυτα στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Όμως, όμως όσον αφορά την ε, ψηφιοποίηση, ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο να το αντιμετωπίζουν ως μια νέα δυνατότητα και όχι μόνο ως μια δυνατότητα σε μια νέα τεχνολογική πλατφόρμα η οποία περιορίζει τις δυνατότητες της. Βεβαίως ε, δεν θέλω να εξαιρέσω και αρνητικά στοιχεία που μπορεί να έχει η ψηφιοποίηση. Ε, δεν πρέπει να ε, θελοτυφλούμε και δεν πρέπει να γνωρούμε πλήρως τις αρνητικές συνέπειες. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που περιλαμβάνει η ειδική έκθεση. Η ειδική έκθεση επισημαίνει ελλείψεις και σημαντικά στοιχεία τα οποία κατά την άποψή μου είναι της αρμοδιότητάς μας. Έχουμε διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, ΦΠΑ, επιβολή δασμών και τα συναφή προβλήματα. Ακριβώς αυτή είναι η τομής στους οποίους εντοπίζουμε τις ε, ελλείψεις και αδυναμίες. Είναι ιδιαίτερα ευτυχές το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι αναγκασμένο τώρα να τρέχει πίσω από τα προβλήματα, διότι έχουμε μία νέα νομική πράξη μέσω της ε, οποίας ε, αναζητάμε ε, και θέλουμε να προσφέρουμε μία λύση για τα προβλήματα. Το 2020 θα τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι νομικές πράξεις και θέλουμε να ελπίζουμε ότι τα υφιστάμενα προβλήματα μπορούν να επιληθούν ή θα μπορέσουν να επιληθούν με αυτές τις ε, νομικές πράξεις. Και έχω κάποια ερωτήματα που θέλουν να απαντηθούν. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Σε σχέση με την ειδική έκθεση κάνατε κάποιες ε, έρευνες και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι οι νέες ε, νομικές πράξεις ε, ετέθησαν σε εφαρμογή πριν από λίγο καιρό και κάποιες θα καθυστερήσουν, θα τεθούν σε εφαρμογή πολύ αργότερα. Από τις έρευνες όμως που κάνατε, ε, πού καταλήξατε, πού βλέπετε να υπάρχουν ε, προβλήματα έτσι ώστε μέχρι το 2021 να μπορούμε να, ε, και να πρέπει κυρίως να συμπληρώσουμε αυτό το νομικό πλαίσιο. Αυτό ήταν το πρώτο μου ερώτημα και το δεύτερο αφορά στις δυνατότητες που έχει το ελεγκτικό συνέδριο ε, σε σχέση ε, με μία αυτοματοποιημένη έρευνα. Πρέπει να το επιδιώξουμε αυτό, δηλαδή ε, κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την επιβολή του ΦΠΑ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υιοθετούμε τις βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες. Ε, στην Ουγγαρία βλέπουμε ότι με την ε, επιβολή του ΦΠΑ επιλύθηκαν πάρα πολλά προβλήματα σε αρκετούς τομείς βλέπουμε ότι έχουμε κλασικές ε, μηχανές καθαρίσεων, τους ε, λογαριασμούς, ε, όλα αυτά μπορούν να εξεταστούν από την Ουγγαρία και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα απάτης. Από την άλλη, πρέπει κάθε μήνα να υπολογίζεται ε, ο ΦΠΑ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όπως αυτό που υπήρχε ε, παλαιότερα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου ε, και του διασυνοριακού ΦΠΑ. Δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόβλημα. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες σχετικά με αυτά τα αυτοματοποιημένα συστήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Λιβιέ Σαστέλ είναι ο σκιώδης εισηγητής μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα πολύ ε, σημαντικό γιατί αυξάνουν ε, χρόνο με το χρόνο οι πωλήσει μέσω ηλεκτρονικού ε, εμπορίου και βεβαίω θα πρέπει όλοι οι εμπορευόμενοι να τα γράφονται για να πληρώνουν τον ΦΠΑ όσο οφείλουν. Ε, και επομένως θα πρέπει να προσέξουμε κυρίως αυτούς που ξεκινούν το εμπόριο από, την, από τρίτες χώρες, πράγμα που δεν διασφαλίζει την καταβολή ΦΠΑ στην ε, χώρα στην οποία καταλήγουν και ε, χρησιμοποιούνται εν τέλει τα ε, προϊόντα. Ε, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε τις αποστολές χαμηλής αξίας απροερχόμενες από τρίτες χώρες. Ε, θα πρέπει να δούμε αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο όμως θα αρχίσει να, να ισχύει από το 2021. Αυτοί που έχουν αναλύσει και από κοντά το θέμα στην στο ελεγκτικό συνέδριο να μας πούν ε, ποιες είναι οι διατάξεις ε, που θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, υλοποιηθούν έτσι ώστε να μην υπάρξει απάτη ΦΠΑ, ποιες είναι οι τεχνολογικές μέθοδοι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η απάτη ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι γεγονός ότι οι φορολογικές αρχές δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι το σωστό ποσό ΦΠΑ θα καταβληθεί εν ευθέτω χρόνο στην ε, αρμόδια χώρα. Άρα ποια είναι τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε συστηματικά να αυξηθεί η διεθνή συνεργασία και η συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών αφενός, αλλά ε, και ε, με οτιδήποτε σχετίζεται με τους εμπορευόμενους που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ganz herzlichen Dank. Äh, Τώρα, από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φερνάντες, η ε, Διευθύντρια, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Oh, sorry. Ε, με συγχωρείτε, πρώτα θα δώσουμε... Είμαι σκιώδη συγκίτρια, λέει η κυρία Κρέτου. δεν μας ενημέρωσε το ΕΛΚ. Πρώτα η σκιώδης και μετά η διευθύντρια, με συγχωρείτε. ναι, λυπάμαι, λέει η Πρόεδρο. Δεν είχαμε ε, λάβει καμία ειδοποίηση, ούτε και το ΕΛΚ δεν μα έδωσε τη σχετική ειδοποίηση. Γι' αυτό λυπούμε αν σα αγνόησα. Η κυρία Κρατσού χωρί. μικρόφωνο. Ωραία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πάρω το λόγο γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για μένα. Ε, πρέπει να σας πω ότι την ε, ε, τελευταία εβδομάδα δούλεψα σχεδόν αποκλειστικά πάνω στο θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε, θα ήθελα να πω και στον εισηγητή κύριο Ντόιτς αλλά και στα αρμόδια εισηγήτρια από το ελεγκτικό συνέδριο να τους πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ε, ξεκινώντας βεβαίως από τη διαπίστωση ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ε, έχει εκρηκτική άνα τον τελευταίο καιρό, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να καταπολεμήσουμε ε, όλες τις παράπλευρες, τα παράπλευρα προβλήματα το 2019 ε, είχαμε 620 εκατομμύρια που χάθηκαν λόγω μη καταβολής των φόρων και βεβαίως η τάση είναι αυξητική από το 1,7 το 2013 έχουμε φτάσει σχεδόν στο 5% το 2019 ε, uh, ο όγκος ε, του ε, εμπορίου και η επίπτωσή του μάλλον στο συνολικό εμπόριο όλο και αυξάνεται όμως και το ποσοστό των ε, των προϊόντων που οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αγοράζουν εκτός των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εδώ ε, θα έπρεπε οι δασμοί ε, και οι φόροι που σχετίζονται με την εισαγωγή να φέρουν ικανοποιητικά, ικανοποιητικούς πόρους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Ντόιτς αναφέρθηκε σε κάποια παραδείγματα τα οποία λειτουργούν καλά, αλλά λυπούμε γιατί πρέπει να πω ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πραγματικότητα ε, φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετική. Δεν έχουμε ούτε καν ε, ε, υπολογισμό των ποσών σχετικά με μη καταβληθέντα ποσά για το ΦΠΑ ή τους τελωνιακούς δασμούς έχουμε έναν γενικό υπολογισμό 5 δις ευρώ απώλειας ανά έτος. I will try shorter. Ε, ε, Κατά την άποψή μου, είναι ανεπαρκής η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μέλων για το θέμα αυτό και ε, ελείπει οπωσδήποτε και η διοικητική συνεργασία μεταξύ χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μεταξύ χωρών Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτων χωρών. Ε, ε, θα πρέπει το Central Liaison Office να έχει μια ειδική μονάδα για το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου Λυπούμε γιατί τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν το Eurofisk ως πλατφόρμα ανταλλαγής ε, πληροφοριών, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική βάση δεδομένων και αν παίξουν όλοι το παιχνίδι οι ευρωπαϊκές χώρες θα γίνει μια πολύ σοβαρή βάση δεδομένων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί ε, το ε, διοικητικό άχθος από τους ώμους των εμπορευομένων και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες στα πλαίσια μιας πραγματικά ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Εγώ είμαι ένθερμη υποστηρίκτρια της ε, δημιουργίας μιας τελωνιακής υπηρεσίας Άλλωστε και ο Επίτροπος Γιωχάνης Χάν ε, στις γραπτές του απαντήσεις ε, απήντησε, ανέφερε ότι θα μελετήσει δεόντως ε, το θέμα της δημιουργίας ενός τέτοιου οργανισμού που θα μπορούσε να αυξήσει τις, τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ε, οργανωθούν όλες οι χώρες ε, σε συνεργασία έτσι ώστε να βρουν ποια είναι τα ασθενή σημεία εισόδου και αυτά τα οποία ε, πιο εύκολα επιτρέπουν την απάτη, ενώ μέχρι τώρα απλώς κυνηγούν αυτούς που έχουν διαπράξει απάτες. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. θα επιτρέψετε και μία συμπληρωματική ερώτηση από την Καταρίνα Κινίτσι. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε και τους ε, ε, προσκεκλημένους μας, το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστούμε τους συγητές και τους και οδησυγητές γιατί το όλο αυτό θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και περίπλοκο. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ γρήγορη, θα τα πω πολύ γρήγορα. Έχω μια ερώτηση να κάνω. Νομίζω ότι είναι Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να εμβαθύνουμε. Η συνάδελφος κυρία Κρεπτή αναφέρθηκε στο σύστημα Eurofiscal Database, ε, αποκεντρωμένο τέτοιο σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις διοικήσεις ε, των κρατών μελών. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό ακριβώς ε, για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Από την έκθεση προκύπτει ότι αυτή η τράπεζα δεδομένων έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Εγώ λοιπόν ε, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι είδους παρεμβάσεις, τι είδους υποστήριξη μπορεί να προσφέρει για να βελτιώσει την ανταλλαγή ε, πληροφοριών, ε, ανταλλαγή πληροφοριών ε, των στοιχείων των τραπεζών δεδομένων για να αποφεύγεται η απάτη. Και εδώ και δύο μικρές διευκρινήσεις θα προσθέσω. Σήμερα γνωρίζουμε ότι από πλευράς όλα δεν υπάρχει απόλυτη πρόσβαση σε αυτό το σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να προσφέρεται στην Όλαφ η πλήρης πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Και κάτι άλλο, ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, πιστεύετε ότι θα μπορεί εκείνη να παρακολουθεί τις απάτες του ΦΠΑ. Έχοντας ε, Κατά όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέπεται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρόσβαση στο Eurofisk για να μπορεί να κάνει ε, σύγκριση των στοιχείων. Και όλοι οι προλαλήσαντες είπαν ότι αυτές οι απάτες προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ganz herzlichen ε, δεν ξέρω πως ξέχασα κάποιον. Αν όχι, κυρία Διευθύντρια, θα δώσω το λόγο σε εσάς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο για την έκθεσή του, την οποία και σημειώνουμε σε ό,τι αφορά τι συστάσει τη. Ε, Σα ευχαριστώ για τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα εδώ. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμφωνούμε με τους ε, σημαντικούς κινδύνους που παραμένουν σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της σωστής ε, ε, παράληψης και συγκέντρωσης των πόρων, ΦΠΑ και δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε διατεθειμένοι και πέραν των νομοθετικών προτάσεων να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη στην πάλη τους κατά της απάτης. Για την Επιτροπή υπό τον Πρόεδρο Γιούγκερ, η καταπολέμηση της απάτης αποτέλεσε μία από τις βασικές της προτεραιότητες. Γι' αυτό και έχουμε προωθήσει μία σειρά νομοθετικών προτάσεων με αυτό τον σκοπό ακριβώς. Θέλουμε μεταξύ άλλων να βελτιώσουμε τη συγκέντρωση πόρων ΦΠΑ, των ε, διαδικτυακών πωλήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών και το καθεξής. Μία από τις βασικές ε, προτάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο το 2018 και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τώρα, γιατί παίρνει τόσο πολύ. Ακριβώς επειδή όλα τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να θεσπίσουν εύρωστα συστήματα πληροφορικά για να διασφαλίσουμε τα δεδομένα και να διευκολύνουμε τους εμπορευομένους να καταβάλουν το ΦΠΑ που τους αναλογεί. Τώρα υπάρχει και μια πρόταση ε, που έχει κατατεθεί από την ε, Κομισιόν, ε, από το Κοινοβούλιο και συζητείται στο Συμβούλιο με μια νέα εργαλειοθήκη για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου από τα κράτη-μέλη η πρόταση θα βοηθήσει τις αρχές να ανταλλάξουν δεδομένα σε σχέση με πληρωμές που έχουν να κάνουν με συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Γι' αυτό και καλούμε το Κοινοβούλιο που τώρα ξεκινά αυτή τη διαδικασία και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις ε, για να υλοποιηθεί η πρόταση το συντομότερο δυνατών. Γιατί θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε έτσι να εντοπίσουμε τους ε, απατεώνες και να αποτρέψουμε τις απάτες. Αυτές οι αλλαγές θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της απάτης, αλλά, όπως αναφέρεται και στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου, και η τεχνολογία μπορεί να διδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και εμείς ε, διερευνούμε και αξιολογούμε μαζί με τα κρατημέλη πιθανές χρήσεις νέων τεχνολογιών για την καταπολέμηση της απάτης. Ήταν και μία από τις ε, συστάσεις στην έκθεση TAX 3, την οποία υιοθετήσαμε. Θα ήθελα επίσης ε, να επισημάνω κάτι που ανέφεραν και οι σκιώδεις τα 5 δις που είπατε ότι χάνονται, εμείς θεωρούμε ότι είναι ακόμα παραπάνω. 7 δις το χρόνο. Και ξέρουμε ότι, πρόκειται για ε, ότι αναπτύσσεται εκθετικά το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτό θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Ε, προσπαθούμε να ασκήσουμε πιέσεις και στα κράτη-μέλη ε, για να αναλάβουν δράσεις προς αυτό το σημείο. Ο κύριος επεσήμανε και το ζήτημα της αυτόματης ε, συλλογής ε, ΦΠΑ. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία εξετάζουμε με τα κάτι μέλη για να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια τέτοια λύση για να διακολύνουμε τέτοιου είδους ίσπραξη σε πραγματικό χρόνο να ενημερώνονται οι αρχές. Τώρα, για τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέσατε. Διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Να υπενθυμίσω ότι και εδώ υπό αυτή την επιτροπή υπήρξε τροποποίηση του κανονισμού για το ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τη διοικητική συνεργασία που θα τεθεί σύντομα σε ισχύ. Ο κανονισμός ενισχύει το ρόλο των κρατών μελών και σε ό,τι φορά τη συνεργασία με τον ε, Όλαφ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ανταλλαγή αυτών των ε, στοιχείων. Με αυτόν τον κανονισμό λοιπόν ενισχύουμε τον ρόλο της Eurofisk και θέλουμε και τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν την υιοθέτηση μέτρων ούτω ώστε η Eurofisk να γίνει ένα πιο πυροδραστικό ε, δίκτυο μεταξύ κρατών μελών. Για τα τελωνία τώρα και τους δασμούς. Ε, συνεργαζόμαστε με κάτι μέλη για να βελτιώσουμε περαιτέρω τους τελειανικούς ελέγχους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κριτήρια οικονομικού κινδύνου και την αξιολόγηση ε, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εμπορευομένων. Αποδεχόμαστε τα όσα είπε το Ελεγκτικό Συνέδριο και έχουμε δημιουργήσει μια νομαλή διαδικασία. Επισκεπτόμαστε όλα τα κρατημέλη για να αξιολογήσουμε το σχετικό αυτό πρόγραμμα και να κάνουμε συστάσεις για την αντιμετώπιση ε, τυχών αδυναμιών. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η διαδικασία. Για τις διεθνείς ε, πτυχές ε, του τηλεανικού σκέλους, στον ΟΣΑ και στον ΠΟΤ έχουν επίσης ενισχυθεί αυτές οι συνεργασίες και εμείς συμμετέχουμε σε αυτά τα βήματα και ασκούμε πιέσεις για την ενίσχυσή τους. Για τον ΦΠΑ, όπως ενδεχομένως έχετε ακούσει, υπάρχει συμφωνία με την Νορβηγία για τη διοικητική συνεργασία που ετέθησε ισχύ πρόσφατα και ήδη έχουμε ωφέλη σε αφορά την καταπολέμηση της απάτης. Αυτή η συμφωνία λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει για να αποτελέσει πρότυπο ενδεχομένω για άλλες τέτοιες συμφωνίες στο μέλλον. Κλείνοντα, θα ήθελα να επισημάνω ότι στις ε, κατευθυντήριες, ε, πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της ε, νεοεκλεγή σα Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται ότι θα ενταθούν οι προσπάθειε καταπολέμηση τη φορολογική απάτη. Φυσικά είναι κάτι το οποίο υφετούμε ω υπηρεσίε τη Κομισιόν και σε ό,τι αφορά τα τελωνία, ανέφερε ότι θα περάσει πλέον η Ελληνική Ένωση σε επόμενο, ανώτερο επίπεδο σε ό,τι αφορά την προστασία της ενιαίας αγοράς και των πολιτών. Εμείς από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να υποβάλουμε νομοθετικέ προτάσει για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν ε, την απάτη, ιδίω στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όμω, παράλληλα, θέλουμε να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη μέσω ε, δικτύων, μέσω ανταλλαγή ε, στοιχείων μεταξύ διοικήσεων για να έχουν τι βέλτιστε πρακτικέ να καταπολεμήσουν την απάτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς ε, πολύ κυρία Διευθύντρια. Επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ έτσι ένα συγκρατημένο σχόλιο. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, κυρίως στο θέμα των κοινωνικών μέσων, θα πρέπει ε, να ομολογήσουμε ότι ακόμα και στη Γερμανία οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να δώσουν κάποια ικανοποιητική απάντηση. Γιατί, διότι δεν υπάρχει ακόμα ε, αρκετή εμπειρία σε επίπεδο οικονομικών υπηρεσιών. Και επειδή η Γερμανία δείχνει να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα των ε, φόρων και της ε, φορολογίας, υποπτεύομαι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα αυτό. Εγώ μία φορά προσπάθησα να ε, διαβάσω λιγάκι προσεκτικά την οδηγία για το ΦΠΑ και πρέπει να σας ομολογήσω ότι ε, σχεδόν άρχισα να αμφισβητώ για την νοημοσύνη μου. Αναγκάστηκα να καταφύγω σε άλλους να μου εξηγήσουν ε, περί τίνος ακριβώς πρόκειται και έτσι δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι επί 14 ολόκληρες μέρες θα προσπαθήσουν να διαβάσουν κάτι όπως το προσπάθησα εγώ για να κατανοήσουν ε, το τι ακριβώς κάνουμε εδώ. Αυτή έτσι είναι μια πολύ συγκρατημένη παρατήρηση. Νομίζω ότι και σε αυτήν την περίπτωση ε, οι πολίτες ε, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταβάλουν φόρο ε, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την νομοθεσία ε, και κατόπιν τούτου ως Επιτροπή Ελέγχου Προεπλογισμών οφείλουμε να μεριμνήσουμε, να εξηγήσουμε τουλάχιστον περί τίνος πρόκειται έτσι ώστε όσοι έχουν καλή τέληση ε, πράγματι να πληρώσουν και οι άλλοι που ε, θέλουν να εξαπατήσουν να συλλαμβάνονται γιατί το 95% που αναφέρεται ως ποσοστό είναι πολύ ψηλό ε, έχουμε λοιπόν πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας και θα καλέσω και τους συντονιστές να το προσέξουν το όλο θέμα γιατί νομίζω ότι το αξίζει τον κόπο το Κοινοβούλιο να προσέξει αυτό το θέμα. Ε, θα θέλαμε και εμείς να μπορούμε να στηρίξουμε το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος επιθυμεί να λάβει το λόγο από πλευράς ευρωβουλευτών. Παρακαλώ, η Κορίνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη προσοχή το θέμα που σχετίζεται με τις επικοινωνίες ε, και με την επικοινωνία γενικότερα. Πραγματικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι κάποια στιγμή άλλωστε. Εγώ έχω δουλέψει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και καμιά φορά πραγματικά μιλάμε με τρόπο δυσνόητο για τον χυψή ε, πολίτη. Θα πρέπει να μάθουμε να μιλάμε με διαφορετικό μορφότυπο ε, και νομίζω ότι και για την καταπολέμηση της απάτης θα πρέπει να καταφέρουμε να μιλήσουμε πιο απλά, πιο εύκολα και στις υπηρεσίες αλλά και απέναντι στους πολίτες γιατί το φαινόμενο είναι πολύ ανησυχητικό. Ε, η Eurostat ε, σε πρόσφατη υπομομέτρηση ε, βρήκε ότι 7 ε, στους 10 πολίτες αισθάνονται ότι υπάρχει απάτη η οποία εν τέλει ζημιώνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης και άρα τον δικό τους προϋπολογισμό. πραγματικά σας ευχαριστώ που θίξατε το θέμα αυτό. Είναι θεμελιώδου σημασίας κατά την άποψή μου. Πολύ ωραία λοιπόν. Ε, θα ήθελα να δώσω πίσω το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις σας, ιδίως προς τον εισηγητή και τους σκιώδης, την κυρία Κρέτσου, την κυρία Κινίτσι και τον κύριο Σούστερ. Θα ήθελα να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα από κοινού, αν μου επιτρέπετε. Η περίοδος ελέγχου κάλυπτε μια περίοδο από την αρχή του 2015 μέχρι τα τέλη του 2018. όπου υπήρχε σχεδόν πλήρης υλοποίηση. Ήδη το 2003 έχει τεθεί σε ισχύ η σχετική απόφαση για τις τρίτες χώρες και οι κανόνες ε, του B2C των υπηρεσιών από ευρωπαϊκές χώρες ε, τέθησε σε ισχύ στις αρχές του 2015. Η πρόταση που επιβλήθη υπό τη δέσμη ηλεκτρονικού εμπορίου στα τέλη του 2017 δεν θα είναι πλήρως εφαρμοστέα μέχρι το 2021, όπως ανέφερε και ο Ταμάς. Έτσι, συνολικός έλεγχος της δέσμης σε ηλεκτρονικού εμπορίου δεν μπορεί να γίνει μέχρι το 2023-2024. Μέχρι τότε θα κάνουμε φυσικά και την απαραίτητη παρακολούθηση. Δεύτερο ερώτημα αφορούσε το σύστημα ίσπραξης. Ναι, εμείς προτείναμε ένα τέτοιο σύστημα και προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει ε, πιθανά κατάλληλα τέτοια συστήματα που θα βασίζονται στις τεχνολογίες. Όμως δεν ήταν σκοπός μας να προσδιορίσουμε περαιτέρω τις τεχνολογίες αυτές. Απλώς καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το διερευνήσει. Τέτοιες πιθανές λύσεις λοιπόν ε, που μπορούν για παράδειγμα να κάνουν χρήση των τεχνολογιών blockchain. διάφορα μέσα πληρωμών που πρέπει να διερευνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τα κράτη-μέλη. μετά τα προβλήματα που ακόμα πρέπει να επιληθούν. Δύο είναι κατά κύριο λόγο. Πρώτον η υποτίμηση και δεύτερον συνεργασία με τρίτες χώρες. Τα έχετε ήδη αναφέρει, αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα. Έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι το 2021. Και οι συστάσεις μας ε, αυτό το στόχο έχουν. Αυτό που ανέφερε η κυρία Κινίτσι για τη Eurofisk. Ναι, πράγματι. Για τον κανονισμό του Συμβουλίου 2018 κάθετος 59, 15 41, πράγματι διευκολύνοντας τη Eurofisk να λαμβάνει στοχευμένες πληροφορίες από τη Europol και από το Γραφείο καταπολέμηση της Απάτης. Υπάρχει λοιπόν αυτό το σύστημα. Πρέπει λοιπόν να το βελτιώσουμε, να προσθέσουμε και νέα στοιχεία για να αυξήσουμε την προσταθεμένη αξία. Ευχαριστώ. Ganz herzlichen Dank. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. κύριε κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω να είμαι πραγματικά λακωνικός. Ε, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως συμφωνούμε όλοι από αυτού ε, και όχι μόνο για λόγους ε, ευγένειας, συμφωνούμε και με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ε, στην συζήτηση προέκυψε ότι όλοι συμφωνούν με ε, την ε, ποιότητα της εργασίας. Ευχαριστούμε την κυρία Ήλτη Κομπαλπέρ και τους συνεργάτες της βεβαίως. Ακούσαμε με προσοχή και την Κομισιόν. Είστε διευθύντρια αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Ε, Κοιτάξτε, στο παρελθόν ε, πραγματικά ε, είχαμε έτσι μια μικρή απογοήτευση όταν ακούγαμε την Κομισιόν. Όμως, στη δική σας ε, περίπτωση πραγματικά βλέπουμε να υπάρχει βούληση για να προχωρήσει το θέμα. Δεν μας απογοητεύσετε καθόλου με αυτά που μας είπατε. Όσον αφορά τους συναδέλφους, οπωσδήποτε θα λάβω υπόψη μου όλες τις παρατηρήσεις σας ε, για την κοινή θέση. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με αυτά που έλεγε πριν από λίγο η Πρόεδρος, δηλαδή ε, κατά την άποψή μου μετά από το 2008-2009, δηλαδή όταν όλοι στην Ευρώπη άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι η κρίση είναι και οικονομική αλλά και ε, έτσι ηθική και δημοσιονομική κλπ. Όλοι τότε ε, τα λάβαμε, ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια ζητήματα, ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις παιδικές ασθένειες ε, ας πούμε ε, και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είναι η φάση της καινοτομίας, η φάση της τεχνολογίας. Ε, χρειαστήκαμε 10 χρόνια και εδώ στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη για να το καταλάβουμε αυτό καλά, ότι πρέπει να προσαρμοστούμε δηλαδή στις νέες τεχνολογίες και στις νέες νέες συνθήκες. Ε, ε, εν όντως, σιγά σιγά εγκαθιδρύσαμε συστήματα ελέγχου των τραπεζικών ε, συστημάτων. Ξέραμε ότι οι τράπεζες ευθύνονται σε μεγάλο μέρος για την κρίση και πολλές τράπεζες στην Ιταλία, στην Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία εστράφησαν προς τα ε, κράτη-μέλη. Δηλαδή, ε, ναι, είδαμε ότι όταν τα πράγματα πάνε καλά οι τράπεζες δεν θέλουν καμία σχέση με το κράτος, όταν αρχίζουν και ζορίζονται τα πράγματα και κυρίως τα οικονομικά, τότε ζητούν και η οικονομική συνδρομή από το κράτος. Είναι σημαντικό, από τη στιγμή που έχει εξελιχθεί μια νέα κατάσταση, να ρυθμιστεί αυτή η νέα κατάσταση. και όσον αφορά ε, τον ανταγωνισμό ε, θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να τον ε, να ρυθμίσουμε ε, και το θέμα του ανταγωνισμού γιατί επηρεάζεται και από τον, το ηλεκτρονικό εμπόριο και από την μη καταβολή του ΦΠΑ από αυτούς που θα έπρεπε να καταβάλουν τον ΦΠΑ είτε αγοράζουν ε, κάτι σοβαρό είτε αγοράζουν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα από το ίντερνετ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, να είναι τόσο απλοί οι κανόνες έτσι ώστε ένας έξυπνος 12χρονος Ευρωπαίος να μπορεί να τους ε, κατανοήσει τους ε, κανόνες αυτούς. Ε, το επίπεδο κατανόησης ε, λοιπόν των οδηγιών ε, θα πρέπει να γίνεται κατανοητό, αντιληπτό από έναν 12χρονο. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να καταλαβαίνει τους κανόνες ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, μας ενδιαφέρει και ένα νέο παιδί να μπορεί να τους καταλάβει τους κανόνες αυτούς. και νομίζω ότι πολλοί μπορεί να η εργασία μας από μια πιο απλουστευμένη διατύπωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το μόνο θέμα που απομένει είναι ε, πώς θα διαμορφώσουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό βέβαια είναι δουλειά των συντονιστών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία το έγγραφο εργασία. Φτάσαμε στο τέλος της ε, ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ όλους και την κυρία Διευθύντρια ε, και τους ε, συναδέλφους. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου 9 μέχρι 12.30 αν δεν κάνω λάθος. Και έτσι λοιπόν η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώνεται οι συντονιστές επιθυμούν η συνεδρίασή τους να ξεκινήσει, ξεκινήσει στις 5 η ώρα και όχι νωρίτερα γιατί κάποιοι συντονιστές βρίσκονται σε άλλες συνεδριάσεις, σε ακροάσεις επιτρόπων ή έχουν και ψηφοφορίες. Δεν μπόρεσαν να έρθουν νωρίτερα. Παρακάλεσαν λοιπόν να ξεκινήσουμε στις 5 ε, η ώρα. 4 ε, και 5 ε, Νοεμβρίου Εκεί ε, θα έχουμε μια κανονική μερίσια διάταξη και νομίζω ότι αυτά είχα να σας πω. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, παρακαλώ έρθετε σε επαφή μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι ε, που θα σας ξαναδώ.